κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας ενημέρωσα την Τετάρτη ότι μια σειρά μελών απέσυραν ε, τις υπογραφές τους σε ό,τι αφορά αυτό το αίτημα. Και έτσι λοιπόν ε, δεν ε, υπήρχαν πλέον αρκετές υπογραφές για το, την πρόταση μορφής αυτής κατά της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άρα αποσύρθηκε στο σύνολό τη. Ο κύριος Σαφάουζερ. Γι' αυτό το ζήτημα. Για το θέμα αυτό. Οι υπογραφές είχαν υποβληθεί, επομένως είχαμε τηρήσει τη διαδικασία και κάποια στιγμή αποσύρθηκαν οι υπογραφές. Αλλά υπάρχει νομικό κενό εδώ και θα ήθελα να ξέρω τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση και γιατί παρά το γεγονός ότι τηρήσαμε τους τύπους, εντάξει, αποσύρθηκαν κάποιες υπογραφές, αλλά όσα είχαν γίνει από πλευράς τυπικής είχαν τηρηθεί. Ε, γιατί λοιπόν ε, δεν δέχεστε την πρόταση μομφής κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι είναι ε, κρίμα που δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε, διότι ε, το ψήφισμα δεν, θα, δεν ήταν δεσμευτικό και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην χάσει την επιρροή του για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ακολουθήσαμε τη διαδικασία του κανονισμού. Όποιος υπογράφει τέτοια αιτήματα ε, μπορεί να αποσύρει την υπογραφή του μέχρι τελευταία στιγμή. Αν αποσύρει την υπογραφή του, καταπίπτει η πρόταση εφόσον ασφαλώς δεν αντικαθίσταται αυτή η υπογραφή από την προτασιμοποίηση σύμφωνα με την άκρη 169 του κανονισμού. Και έτσι λοιπόν δεν θεωρήθηκε ότι υπήρχαν επαρκείς υπογραφές και έτσι κατέπεσε λοιπόν η πρόταση μόμφης. Σας ενημερώσαμε λοιπόν και εσάς και όλους τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές προκειμένου να ξέρετε ότι δεν αντικαταστάθηκαν υπογραφές. Και γι' αυτό λοιπόν σας αποστέλαμε τις σχετικές πληροφορίες στις